Ε, Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Ξεκινάμε μάλιστα. Θα ήθελα να ζητήσω στα μέλη του κοινού που έρχονται όλο και πιο πολυπληθείς συνεδρία της Επιτροπής Προϋπολογισμών να κάνουν ησυχία. Καθυστερήσαμε γιατί κράτησε λίγο περισσότερο συνεδρία των συντονιστών, ήταν ιδιαίτερα πεφορτωμένη η ημερησία διαταξή του και εμείς έχουμε πολλά σημεία στην ημερησία διαταξή, θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Είναι πέμπτη απόγευμα μετά από μήνυ ολομέλεια. Όλοι θέλουμε να ξαναγυρίσουμε στους εκλογέ μα. Σα παρακαλώ, λίγη ησυχία. Είδατε την ημερησία διάταξη, αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Εγκρίνεται η ημερησία διάταξη. Έχετε στο φάκελό σας το έγκυρο έγγραφο έντυπο Κόμπιου News της ανακοινώσεις του Προέδρου. Δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών Ναι, ναι, όχι, συγγνώμη. Ανακοινώσει έχω να σας πω κάτι. Μου λένε ότι λόγω της παράτασης της Ολομέλειας η τσεχική καμπίνα θα εργαστεί μόνο από τις τέσσερις Συγγνώμη από τους τσέχους συναδέλφους. Σε ό,τι αφορά το 3, την έγκριση των πρακτικών, ως ήθιστε θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά εάν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης δεν εγερθούν αντιρρήσεις ή ενστάσεις. Σας προτείνω να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία, στον χρόνο ψηφοφορία, το σημείο 10 δηλαδή, την έκθεση της Ναντέσκα, Ναντέστα Νέινσκι για τα κριτήρια, τη διεύρυνση, τις πολιτικέ και τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Voilà, vous avez votre liste de vote. Λοιπόν, έχουμε τον κατάλογο ψηφοφορία και σα έχει διανεμηθεί και μια προφορική τροπολογία υπαριθμών 6 που θα παρουσιάσει την κατάλληλη στιγμή η εισηγήτρια όταν ψηφίζουμε την τροπολογία υπαριθμών 6. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ε, είσαστε όλοι έτοιμοι, έχετε τι κάρτε σα, ε, του κατάλογου για την ψηφοφορία, τα έχετε όλα. Ο κύριος Ρικέξ έχασε την κάρτα του. και ο κύριος Καλφίν. Εντάξει, τότε αλληλοξιδετερώνονται. Στην Βουλή των Κοινοτήτων έτσι γίνεται. Ξεκινάμε παράγραφος ένα Συμβιβαστική τροπολογία Α. Ψήφι υπέρ. υπέρ. Συμβαστική Α. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Καλύπτεται. Καλύπτεται. Εν μέρη από τη συμβαστική α, αν εγκρίνουμε και την ε, συμβαστική β, τότε καλύπτεται πλήρως. Περνάμε στην τροπολογία 4. Λίγη ησυχία παρακαλώ, τροπολογία 4. Ο εισηγητής είναι υπέρ, η εισηγήτρια υπέρ, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3, Μέλτσερ, <clears throat> συμβατή, ο εισηγητής είναι κατά, ψήφι υπέρ. Κανείς. Δύο. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5, Παξά, συμβατή, η εισηγήτρια είναι υπέρ, ψήφι υπέρ. Κατά. αποχές μία πλειοψηφία κατά του ΕΛΚ απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Προφορική τροποποίηση της εισηγήτριας που έχει ε, διανεμηθεί. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. <clears throat> Νέσδα. Ναι, Θέλουμε να κατεβάσουμε μια τροπολογία προφορική. Τι που θα πρέπει να δει ε, ποιοι είναι δικαιούχοι ε, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτή την ε, πτώση της χρηματοδότησης το οποίο να σημαίνει ότι η, η αρρωγή αυτή που θα ενισχύσει κάθε χώρα στο ΑΕΠ δεν πρόκειται να μειώσει σχετικά ακόμα και τον ε, παρονομαστή για κάθε χώρα δικαιούχο και σε αυτή την περίπτωση το ποσοστό της χρηματοδότησης ανά ΑΕΠ, ούτως ώστε να καλυφθούν τα συστημικές βελτιώσεις από πλευράς θεσμικών αλλαγών. Είναι προφορική τροπολογία. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να αντικαταστήσουμε αυτό το κομμάτι με εκεί που λέει σορευτική αύξηση για την περίοδο το 2007-2013 για την κάθε χώρα τόσο από η Κροατία αύξηση 10% με την αναλογία της συνολικής αρρωγής IPA που δεν θα πρέπει να μειωθεί ακόμα και αν αυτό ο παρονομαστή κάθε χώρα δικαιούχου πρόκειται να έχει αυξηθεί σωρευτικά σε πραγματικού όρου κατά την περίοδο 2007-2013. Επίση έτσι θα πρέπει να απαλληφθεί η υποσημείωση εκείνη η οποία λέει οι ίδιες εκτιμήσεις με στοιχεία της Γενικής Διεθνής του και προβλέψεις για τις υποψήφιες χώρε και επίσης να υπάρχουν κάποιες προβλέψεις που θα βασίζονται σε κάποιες εκθέσεις κάποιας ανεξαρτήτου ε, εταιρεία, κάποιο ανεξαρτήτου φορέα προβλέψεων. Έχετε το λόγο διαδικαστικό, πρόεδρε. Είναι δύσκολο να τοποθετηθούμε πάνω σε αυτή την ε, προφορική τροπολογία, γιατί μας ήρθαν τη 12η ώρα, τώρα μόλις θα δουλεύει συμφορία, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε γραμμή. Τι να σας πω, δεν, δεν, δεν, δεν ξέρω πού να βασιστώ για να συμφωνήσω ή όχι. Κύριε Φάρμ, εγώ φταίω, εγώ φταίω. Γιατί ήθελα να αλλάξω το αρχικό κείμενο Αντές σε ευχαριστούμε που το ότι μας γιατί το αρχικό κείμενο ήταν δυσνόητο. Αυτό είναι πολύ σαφές. Το τόσο η ουσία δεν αλλάζει. Ωραία, θέτω σε ψηφοφορία λοιπόν την τροπολογία. Τροπολογία 6 με την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. φιλελεύθερη και κάποιοι άλλοι αποχές. Και δύο, συνάδελφοι, δύο Ισπανοί συνάδελφοι απέχουν. Υπάρχει πάντως μια πλειοψηφία. Α, ναι, και, και, α, και Πολωνός και Πολωνός. Και Ισπανό Ισπανοπολωνική είναι η Σες. Α, oui, non, α, και Γαλλική, Γάλλο-Πολωνο-Ισπανική. <laughs> You want to check? Okay, okay, okay, okay, okay. We check, we check. Να γίνεται τόσο έλεγχος. Ναι, ναι, ναι. Ελέγχουμε, ελέγχουμε. Τροπολογία προφορική. Allez, votez, votez, votez, votez. Voilà. Ψηφίζουμε. Κάποιος δεν έχει ψηφίσει. Πέρασε. Vote clos. 12 pour, 10 contre, 4 abstentions. 12-10 με 4 αποχές. Monsieur Riquet s'est abstenu. il s'est abstenu. Ε, Donc, une euh, courte majorité. Άρα έχουμε μια μικρή πλειοψηφία. Τροπολογία του 7 του κυρίου Μέλτσερ είναι κατά ο συγκητής, ε, Ποιο είναι υπέρ, Σα ευχαριστώ. Ε, απορρίπτεται 8. Πάξα. Είναι κατά ο συγγητή. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ναι. Φάρν. Συμβατή. Είναι κατά ο εισηγητής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Είναι η πλειοψηφία κατά και απορρίπτωται. Οκτώ. Φέρν. Είναι υπέρ ο εισηγητής. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Εγκρίνεται. Δέκα του εισηγητού. Συμβατή. είναι κατά. Τι είναι υπέρ. Υπέρ. Πριν ο πρόεδρος. Κατά λέει τώρα. Ευχαριστώ αποχές. Υπέρ είναι η πλειοψηφία. 12. Νίτσκι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική Β κεφαλαίου του εισηγητού. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επομένως, η υπαριθμόν δύο τροπολογία καλύπτεται από το α και β συμβαστικές. Τώρα έχουμε την 13. 13 ε, καλύπτεται, 14 νίσχυ, ναι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 φέρν υπέρ ο υπέρ, κατά. Ομόφωνα εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Σας προτείνω ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε και είστε υπέρ και εσείς. Πέρα ψηφοφορίας ψήφισαν όλοι. 23 υπέρ. Δύο κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια. Ναι, ναι, το αξίζουν ε, χειροκροτήματα. Και φυσικά χειροφίλημα. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο σημείο παριθμών 11. Υπάρχει εδώ μία μεταφορά πίστοσης.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 Στις 8 Μαΐου στη συνεδρίασή μας είχα παρουσιάσει τα στοιχεία <clears throat> για αυτή τη μεταφορά, τώρα θα την ψηφίσουμε. Είναι κάτι που χρειάζεται για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, πρέπει να γίνει αυτό πριν από το καλοκαίρι. Υπάρχουν λοιπόν κάποια στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση του προγράμματος Χρειάζονται λοιπόν να γίνονται αυτές οι πληρωμές πριν από το καλοκαίρι. Επομένως θα έχουμε αυτές τις ε, που προτείνει η Κομισιόν. Ο Σαλβαδόρ Γαρία. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, κάνει μια θέληση να εμποδίσω το χρονοδιάγραμμα πληρωμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα πλαίσιο. Είχαμε ζητήσει όμως πρόσθετες πληροφορίες για την κατάσταση στην οποία βρισκόνται τα προγράμματα <clears throat> τα οποία δεν είχαν εφαρμοστεί πλήρως και τα οποία οδήγησαν σε αυτήν την ε, ε, υπερβολική ποσότητα πληρωμών σε σχέση με τις ανάγκες. Βλέπω τώρα ότι στο επεξηγητικό σημείωμα δεν μας δίνονται οι πληροφορίες αυτές για τα προγράμματα και αυτό νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να ξέρουμε σε ποια προγράμματα έχει γίνει η υπερβολική αυτή οι υπερβολικές αυτές πληρωμές γιατί όταν εμείς είπαμε ότι θα πρέπει να ανακτήσουμε κάποιες πιστώσεις που προέρχονται από άλλες σε άλλες γραμμές του προϋπολογισμού όπως η Γεωργία είχαμε ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες για να έχουμε καλή, μια καλή εικόνα για να ξέρουμε τι ακριβώς δεν πήγε καλά στην διαδικασία εφαρμογής. Γιατί πρέπει πάντα να προσαρμόζουμε τους πόρους στις ε, αναγκαιότητες και αυτή είναι μια σαφής περίπτωση που δεν υπήρξε αντιστοιχεία των πόρων με τις ανάγκες. Αν θέλει η συγγύτρια να ψηφίσουμε για λόγους κατεπήγοντος, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι εμείς ως Επιτροπή Προϋπολογισμού πρέπει να έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες. Ευχαριστώ κύριο Σάλβαρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω πως μέχρι την τελευταία πρόταση υπέθετα πως ε, ο κύριος Γκαρίγκα θα ζητούσε μετά να καταψηφίσουμε αυτή την ε, μεταφορά. Να σας πω κάτι ουσιαστικό. Εάν δεν έχουμε τις ε, πληροφορίες, γιατί θα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Για μένα θα έπρεπε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Για μένα δεν υπάρχει θεωρώ τίποτα χειρότερο από το να πηγαίνουν κονδύλια από τον τομέα σε ενεργειακά δίκτυα, ε, διαφορετικές πηγές ενέργειας, πρωτοβουλίες ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να αφαιρούνται όταν σε κάθε χώρα της Ευρώπης λέμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την ενέργεια, εναλλακτικέ ενέργειες κτλ. Και στη δικιά μου. Οπότε, ανεξαρτήτως της ε, δυνατότητας και του κατεπήγοντος ίσως αν και αναρωτιέμαι για την εξάντληση του αποθέματος. Αλλά ακόμα και μόνο το, βήμα, το μήνυμα που στέλνουμε, δηλαδή παίρνουμε τα λεφτά από τα μελλοντικά δίκτυα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τι πάμε στη γεωργία, είναι μοιραίο λάθος. και θα ήθελα να παραμείνουν αυτά εκεί πέρα ως μήνυμα στα κράτη-μέλη ότι αν δεν τα χρησιμοποιήσετε αυτά τα λεφτά εξαφανίζονται αλλά είναι δική σας ευθύνη. Γιατί το μήνυμα ε, νομίζω που θα στείλουμε αλλιώ, ε, ειδικά σε αυτούς τους χερούς είναι πραγματικά μοιραίο. Ε, Ευχαριστώ. Εγώ από προσωπική άποψη δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση μετά τη χθεσινή συνεδρία Είχαμε αναφερθεί προηγουμένω στη συνεδρία των συντονιστών ποια ήταν τα διδάγματα που προήλθαν από τη συνάντηση σε σχέση με τα κριτήρια πληρωμών όπου υπήρξε μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής Προϋπολογισμών με τον Τζορς Λάιον και μια αντιπροσωπεία τη Κομισιόν με επικεφαλή στο Γενικό Διευθυντή προπολογισμών για να δούμε ακριβώ πόσο είχαν εκταμιευθεί τα κονδύλια, αν υπήρχαν καθυστερήσει και γιατί. Φαίνεται ότι το θέμα αυτό δεν αναφέρθηκε χθε ή τουλάχιστον αναφέρθηκε επαρκώς. Μου λένε ότι η τουλαχιστον αναφερθηκε επαρκώ. μου χρονική στιγμή για την Επιτροπή προπολογισμών είναι η 1η Ιουνίου. Εάν λοιπόν τότε υπάρχουν κάποιες πολιτικές ομάδες οι οποίες δεν έχουν πλήρη πληροφόρηση. Έχουμε κάθε δικαίωμα να αναβάλουμε την ε, ψηφοφορία για τη μας 30 και 31 Μαΐου. Νιώθετε λοιπόν ε, σύμφωνοι με αυτό και η συγκέντρια. Ναι, ναι, ναι βέβαια. Δεν υπάρχει πρόβλημα, όσε πιο πολλέ πληροφορίε έχουμε, τόσο καλύτερα θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με καλύτερη γαλήνη. Θα χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο που έχουμε. Αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα στα σημεία που μα έχει δώσει ήδη η Κομισιόν. Υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία σε αυτά που μα έχει ήδη δώσει υπό μορφή εγγράφων η Κομισιόν. Πολύ καλά, λέει ο πρόεδρο. Μα μιλάμε για χοντρά λεφτά. Είναι σημαντική αυτή η μεταφορά πιστώσεων από ποσοτική άποψη και όπως και άλλοι συνάδελφοι και εγώ κάπως νιώθω άσχημα όταν κατανοώ ότι τρία χρόνια μετά την εκκίνηση αυτού του προγράμματος που κάλυπτε 100 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν σε ένα πακέτο 30 δισεκατομμύριων ευρώ 30 δισεκατομμύρια από την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 100 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό. Όλα αυτά ήταν στοιχεία ενός συνολικού σχεδίου ανάκαμψης που σε βασικό επίπεδο ε, χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς σε επίπεδο 300-500 χιλίων δισεκατομμύριων. Ε, τρία χρόνια μετά και όταν η χώρα μας είναι όταν οι χώρες μας είναι σε κατάσταση ύφεση πολλές φορές και υπάρχουν όλα αυτά τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια που δεν έχουν εκταμιευθεί, αυτό θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Έχουμε ένα μικρό προπολογισμό. Προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε όσο δυνατό περισσότερο τις καινοτόμε πολιτικές, τις ε, στοχευμένες επενδύσεις για να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη <clears throat> και την τόνωση της ανάπτυξης. Και όταν θέλησαμε να το κάνουμε αυτό πρόσφατα, σε τομεί που όπω αναφέρει ο κύριο Άλβαρο, Φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες, υπάρχουν πολιτικές προτεραιότητες σε όλα τα κράτη-μέλη. Εκεί δεν τα χρησιμοποιούμε τα ποσά αυτά. Όλα αυτά είναι παράδοξα. Σας προτείνω, συμφωνώντας με την εισηγήτρια και επί τη βάση της προτάσεως πολλών μελών, να αναβάλουμε αυτή την ψηφοφορία για την επόμενη μας συνεδρίαση στις 31 Μαΐου. Και εντωμεταξύ θα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις ε, πληροφορίες που θα έχουμε στα χέρια μας, μεταξύ των οποίων και αυτές από την Εκτελεστική Επιτροπή. 12. Ο κύριος Φερνάντες δεν έχει έρθει, διότι δεν υπάρχει καμία αίτηση μεταφοράς πιστώσεων. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στο σημείο 4, που είναι ο προπολογισμό του 2013 και η εντολή για τον τριμερή διάλογο. Κύριε Λαβία. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ενώ εμείς συζητάμε τα θέματα του προϋπολογισμού για το 2013, λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα, διότι συγχρόνως καθορίζονται οι προτεραιότητες για την χρήση των πόρων που δυστυχώς είναι περιορισμένοι λόγω της κρίσης. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό τη στιγμή που θα πρέπει εμείς να καθορίσουμε την εντολή για το Κοινοβούλιο σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2013, γιατί είναι προφανές ότι θα είναι η δική μας θέση ως Επιτροπής Προϋπολογισμού ως αντίδραση στην αρχική πρόταση της Κομισιόν που θα αποτελέσει θέση του Κοινοβουλίου. Εδώ θα ήθελα να πω ότι σε μια περίοδο κρίσης όπως αυτή που διατρέχει τώρα η Ευρώπη, η πρόταση η οποία θα προέλθει από το Κοινοβούλιο θα πρέπει να σέβεται ιδιαίτερα τις συνθήκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Προφανώς δεν μπορεί να έρθει σε σύγκρουση με το οικονομικό κλίμα βαθιάς λιτότητος που αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν μετά από τις συναντήσεις που έκανα με τους εκπροσώπους των επιμέρους επιτροπών του Κοινοβουλίου, εγώ ζήτησα από όλους τους συνάδελφους στις επιμέρους επιτροπές να εκφράσουν τις πολιτικές τους προτεραιότητες μέσα στα πλαίσια της ε, συνολικής στρατηγικής που είχαμε αναφέρει στις κατευθυντήρες γραμμές, δηλαδή ανάπτυξη ε, και θέσεις απασχόλησης ιδίως για τους νέους. Νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους με το να περικόψουμε εφόσον αυτό είναι απαραίτητο ή αναθεωρώντας ορισμένα προγράμματα τα οποία δεν εντάσσονται σε αυτή τη συνολική στρατηγική αλλά τα οποία έχουν και περιορισμένο επίπεδο απορρόφησης. Επί της βάσης αυτής λοιπόν εγώ έχω βασίσει το σχέδιο για την εντολή του τριγωνικού διαλόγου που έχω αποστείλει χθε σε όλου του συναδέλφου μέσω τη γραμματεία. Υπάρχουν φυσικά και κάποια γενικά ζητήματα για τα οποία εμεί είμαστε υποχρεωμένοι να συζητήσουμε και τα οποία εξ, ε, ε, αφορούν την πρόταση της Κομισιόν σε σχέση με τις ε, πιστώσεις υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών και επίσης αφορούν ορισμένα συγκεκριμένα θέματα. Να σταθούμε καταρχήν στις πιστώσεις υποχρεώσεων που εκφράζουν πάνω απ' όλα τις πολιτικές μας προτεραιότητες και που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χρησιμοποιήσει αυτές τις πιστώσεις για να καταδείξει ποια είναι η ιεράρχηση των προτεραιότητων του σε σχέση με τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα βρισκόμαστε σε μια στιγμή κρίσης με ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο ραλ, δηλαδή υπολοιμάτων από το παρελθόν, πιστώσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί. Δεν μπορούμε μέσα σε μια κατάσταση που το προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ενισχυθεί, η Κομισιόν είχε προτείνει να παγώσουμε τι πιστώσει απασχόληση. Δηλαδή να περιορίσουμε την αύξηση των πιστώσεων υποχρεώσεων μόνο στο επίπεδο του πληθωρισμού, που είναι 2%. Αυτό είναι μια πολιτική, όπω σα λέω, επιλογή, μια στεναρή πολιτική επιλογή, που πιστεύω ότι θα πρέπει να την ελέγξουμε στη συζήτηση που έχουμε να κάνουμε στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου, γιατί μια τέτοια θέση σημαίνει ότι είναι και πάγωμα των προοπτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ είμαι πεπισμένο αντίθετα ότι για να μπορέσουμε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή από την κρίση αυτή της Ευρώπης, για να έχουμε μια διέξοδο από την κρίση, χρειαζόμαστε περισσότερο και όχι λιγότερη Ευρώπη. Και από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια σαφής ανάγκη να καλύψουμε τις πιστώσεις πληρωμών που απαιτούνται. Εδώ έχουμε κάνει μια εποπτεία, μια διαδικασία εποπτική για τις πιστώσεις που χρειάζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγινε σαφές ότι πρέπει να <clears throat> προχωρήσουμε σε πληρωμές σε σχέση με υποχρεώσεις που έχουν ήδη συναυτεί. Η Κομισιόν λοιπόν απεδέχθη αυτό το οποίο είχαμε πει εμείς στις κατευθυντήρες γραμμές μέσω της αίτησης που είχαμε ε, καταθέσει για ένα ρεαλιστικό αλλά και υπεύθυνο προϋπολογισμό. Η πρόταση Κομισιό λοιπόν αποδέχεται αυτά που ζήτησε το Κοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι οι προβλέψεις για τον προϋπολογισμό της Κομισιόν θα είναι επαρκείς για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες. Είδαμε χθε ότι οι προβλέψεις της Κομισιόν λαμβάνουν υπόψη και έχουν και πολιτική στάθμιση σε σχέση με τις ανάγκες, οι οποίες φυσικά είναι πάντα μεγαλύτερες. Όλα αυτά θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε περαιτέρω επαλήθευση μέσα στη διάρκεια του 2012 για το ρυθμό εκταμίευσης των, πιστώτων, των πιστώσεων ε, πληρωμών, ώστε να μην υπάρξει μεταφορά αναγκών πληρωμών από το 2012 στο 2013. Θα πρέπει να αποφύγουμε το 2013 να παραμένουν ακόμα <clears throat> υποχρεώσεις που δεν έχουν οδηγήσει σε πληρωμές και να μεταφέρονται εσαΐ e στον επόμενο χρόνο αυτές οι πιστώσεις. Σε σχέση τώρα με συγκεκριμένες θέσεις του προϋπολογισμού, έχουμε διατυπώσει ορισμένε προτεραιότητες και έχουμε καταδείξει και ποια είναι τα βασικά στοιχεία στο σχέδιο της εντολής για τον τριγωνικό διάλογο. Στην κατηγορία 1α, 4,1 για αύξηση για τις πιστώσεις υποχρεώσεων, 17,8 πιστώσεις πληρωμών. Αυτή είναι η πρόταση της Κομισιόν. Εδώ έχουμε τη μεγαλύτερη ε, συγκέντρωση πιστώσεων υποχρεώσεων, γιατί εκεί περιλαμβάνονται και οι πολιτικές ενέργειες για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης και καταδεικνύουν πλήρως την θέση του Κοινοβουλίου και υποστηρίζουν τις δικές μας προτεραιότητες. Το επίπεδο πληρωμών θα πρέπει να συμβιβαστεί με αυτό που είναι απαραίτητο. Μια ρεαλιστική λοιπόν εκτίμηση είναι απαραίτητη για να καλύψουμε και το κόστος των ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία φτάνουν στο τέλος τους. Επίσης αναγνωρίζουμε το ρόλο που δίνει η Κομισιόν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως κινητήριου μοχλού για την ανάπτυξη και επίσης την διευκόλυνση για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πιστώσεις. Τα επενδυτικά αυτά μέτρα ε, έχουν αυξήσει τη χρηματοδότηση σε σχετικούς όρους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δυστυχώς, η Εποπτική Αρχή και κάποια άλλα προγράμματα δεν έχουν πάρει την απαραίτητη χρηματοδότηση για να μπορέσουν οι φορείς αυτοί να καλύψουν τα, τα εγχειρήματα τα οποία πρέπει να υποστηρίξουν. Να σας υπενθυμίσω επίση ότι υπάρχουν εγχωρισμένα προγράμματα όπως είναι η διαβίου εκπαίδευση η οποία έχει λειτουργήσει πολύ καλά σε επίπεδο εκταμίευσης έχει και τα διευρωπαϊκά δίκτυα που έχουν στρατηγικό χαρακτήρα έχουν αντιμετωπιστεί με θετικό τρόπο από την Κομισιόν. υπάρχει ένα χωριστό κεφάλαιο σε σχέση με το σχέδιο ΙΤΕΡ για το οποίο δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Η Κομισιόν προβλέπει να χρηματοδοτήσουμε 360 εκατομμύρια βάσει της συμφωνίας του περασμένου Νοέμβρη με την επανανάπτυξη κοντιλίων από ορισμένες άλλες γραμμές του προπορισμού, κυρίως τις διοικητικές γραμμές, γραμμές διοικητικών δαπανών του 7ου προγράμματος πλαίσιου. Εμείς θέλουμε όμως να ελέγξουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες μιας τέτοιας αναδιάταξης. Μας φαίνεται ότι είναι απαραίτητο, όπως κάναμε και για τη διάλογο, το Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει πλήρως όλα τα εργαλεία τα οποία, τα οποία είναι απαραίτητα για το δημοσιονομικό κανονισμό στην τριμερή συμφωνία των δύο θεσμικών οργάνων. Έτσι συμφωνήσαμε στην, συνδια... στην ε, πέρσι. Για την κατηγορία 1β, εμείς έχουμε εκφράσει την ανησυχία μας για την κατάσταση των πληρωμών στον τομέα αυτό. Υπενθυμίζουμε ότι η Κομισιόν δεν μπόρεσε να πληρώσει 11 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 2010 που αφορούσαν δισεκατομμύρια συγγνώμη, αφορούσαν θεμητές ε, αιτήσει πληρωμών των κρατών μέλων και έχουν μεταφερθεί ένα τμήμα από αυτά το 2000-2003. Θεωρούμε επίση ότι το επίπεδο των πληρωμών είναι ένα πρώτο και χρήσιμο βήμα για να προσαρμοστούμε στις ανάγκες αυτής της κατηγορίας. Κατηγορία 2. Εδώ υπάρχει μια αύξηση όπως προτείνει η Κομισιόν γιατί φτάνουμε στο τέλος του Ταμείου για τη Σάκχαρη και επίσης μια σημαντική αύξηση των κονδυλίων για τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και για την, ε, το phasing in για τις άμεσες πυρομές και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να υπάρξει μια αύξηση για τα κονδύλια. Θεωρώ ότι είναι θετική πρόταση της Κομισιόν να διατηρήσει την χρηματοδότηση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής ενώ θα πρέπει να συμπεριληφθεί εδώ και η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την κατηγορία 3α όπου αυξάνουν κατά 8% επιστώσεις υποχρεώσεων 1,8% σε σχέση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό και 11% επιστώσεις ε, πληρωμών θεωρούμε ότι όλα αυτά πρέπει να συνάδουν με τις ε, αυξανόμενες Φιλοδοξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα τη ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Ο αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματο που δημιουργεί τόσα πολλά προβλήματα στην οικονομία μα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει επίση να αντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανάστευση. Υπάρχουν κάποια προβλήματα ακόμα υπό για ορισμένε γραμμέ του προπολογισμού και γι' αυτό είναι απαραίτητο να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι που έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. 3β. Ξέρετε όλοι ότι είναι το πιο μικρό, η πιο μικρή υποκατηγορία και εδώ έχουμε μια μικρή μείωση στις πιστώσεις πληρωμών και πιστώσεις ε, υποχρεώσεων. Η Κομισιόν έχει προτείνει την ενίσχυση του προγράμματος νεότητας σε δράση που έδειξε πολύ καλή απορρόφηση πόρων και επίσης έχει πολλές δυνατότητε να προκαλέσει θετικά αποτελέσματα. Χρειάζεται επίσης να υπάρξει μια προσπάθεια να μειωθεί το χάσμα επικοινωνίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των πολιτών. Ένα χάσμα το οποίο πρέπει να καλυφθεί ώστε να έχουμε ένα μεγαλύτερο επίπεδο συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές και ιδίως στην ευρωπαϊκή στην ευρωπαϊκή προεκλογική Εξατία που ελπίζουμε ότι θα έχει υψηλότερο επίπεδο συμμετοχή από ό,τι στο παρελθόν. Κατηγορία 4 είναι μια πάρα πολύ λεπτή κατηγορία, πολύ ευαίσθητη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. όπω ξέρετε, πολλέ φορέ τα τελευταία χρόνια έχουμε παρέμβει και έχουμε τροποποιήσει την πρόταση της Κομισιόν. Η πρόταση είναι 0,7% στις πιστώσεις υποχρεώσεων, 5,1% στις πιστώσεις πληρωμών. Υπάρχει λοιπόν μια σημαντική αύξηση εδώ 272 εκατομμυρίων για το προτινόμενο περιθώριο λόγω θεμάτων που έχουν να κάνουν με το DCI, την προενταξιακή ε, υποστήριξη κτλ. Η Κομισιόν θα πρέπει να μας δώσει όμως εξηγήσει στον τριγωνικό διάλογο για να εξηγήσει γιατί μειώνονται συνολικά οι πόροι προς τα κάτω γιατί αυτό μπορεί να είναι κάτι το κατανοούμε σε περιπτώσεις οι οποίες είχαν υποαπορρόφηση, αλλά δεν θέλουμε να δεχτούμε α, ορισμένες αυθαίρετες περικοπές για την πρωταξιακή στρατηγική. Κατηγορία 5. 2,8 ε, είναι η αύξηση χωρίς να ληφθεί υπόψη η Κροατία. <clears throat> Όλα αυτά είναι ε, αποτέλεσμα συμβατικών υποχρεώσεων που έχουν συναυθεί από τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται λοιπόν να συνεχίσουν οι προσπάθειες για την εδραίωση του διοικητικού προϋπολογισμού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί παρά να υποστηρίξει μια τέτοια προσπάθεια τη στιγμή που βρισκόμαστε σε φάση κρίσης. Νομίζω ότι για τις αποκεντρωμένους φορείς θα πρέπει να πω περισσότερα πράγματα, γιατί το γενικό επίπεδο 748 εκατομμύριων ευρώ για τους αποκεντρωμένους φορείς λόγω του phasing in 7 νέων φορέων που χρειάζονται κονδύλια για να ξεκινήσουν τις δραστηριότητες τους. Εδώ έχουμε εκφράσει κάποιες ανησυχίες γιατί για πρώτη φορά η Κομισιόν έχει περιορίσει την χρηματοδότηση κατά 44 εκατομμύρια ορισμένων φορέων που ήταν ήδη μέσα στα πλαίσια των προτεραιοτήτων μας. Δεν μπορούν όμως οι πόροι των αποκεντρωμένων φορέων να θεωρούν ότι είναι καθαρά διοικητικές δαπάνες, διότι συμβάλλουν με ουσιαστικό τρόπο οι αποκεντρωμένοι φορείς στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ευχαριστώ. Merci de cette présentation très claire et très synthétique, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τόσο σαφή σας ε, εισήγηση. Ε, έχουμε πάρα πολλούς γνωστούς στο λόγο και ο πρώτος πρώτο του η κυρία Γκουαρδιά Θάμπαλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο το οποίο θα ήθελα να σας ε, αναφέρω είναι συγχαρητήρια προς τον κύριο Λαδία. Διότι νομίζω ότι αυτή η έκθεση που απευθύνεται και θα καταλήξει στο ε, τριμερή διάλογο νομίζω ότι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που είχαμε διότι κρατά μια πορεία που θεωρούμε ότι είναι αυτή που θέλουμε να κρατήσουμε σαν ρότα για αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις για το 2013. Είναι λοιπόν κάποια συγκεκριμένα σημεία και ε, θα εξετάσουμε όταν έρθει η ώρα τις ε, τροπολογίες γενικά μέσα στο ίδιο μήκος κύματος όσον αφορά την διαπραγματευτική εντολή εδώ που τονίζει ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα για εξυγίανση των δημιουργικών αλλά επίσης και εκεί που σχολιάζει το ότι χρειάζεται να υπάρχουν επενδύσεις για να φτάσουμε, για να φτάσουμε σε ανάπτυξη. Και όλα αυτά πέραν της τάξης μεγέθους του ε, προϋπολογισμού... Επίσης το ίδιο αφορούν τις ε, πληρωμές μας γιατί διστάζουμε σε σχέση με αυτήν την πρόταση του, του Συμβουλίου για περικοπή στις πληρωμές κάτι το οποίο θα το δεχτούμε ποτέ. Και επίσης και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι πάρα πολύ καλά τα έργα πληρωμές η Επιτροπή. Τώρα όσον αφορά και συγκεκριμένα θέματα ε, εκεί που αναφερόμεθα στην προσχώρηση της Κροατίας, αναφερόμεθα επίσης και ε, στην, στην γενικότερη, στο γενικότερο τμήμα της εντολής και όχι στο κομμάτι της εντολής που αφορά την τρίτη, την τρίτη κατηγορία, το τρίτο κεφάλαιο, γιατί θα γίνει από τον Ιούλιο πλήρε μέλο η Κροατία και οπότε αυτή η υπόθεση τη συγχρηματοδότηση θα πρέπει να ξεκαθαριστεί περισσότερο. Σε γενικές γραμμές, πέραν του, του ότι καταρχήν ε, νομίζω ότι έχουμε κάποιες ε, αυξήσεις ε, όσον αφορά την πρόταση, σε σχέση με την πρόταση του 2013, εάν κάτσουμε και συγκρίνουμε αυτά σε σχέση με τον προγραμματισμό θα, δούμε ότι δεν είναι και τόσο μεγάλες αυτές οι αυξήσεις γι' αυτό και τα τονίζουμε αυτά τα σημεία. Όσον αφορά τώρα την καταπολέμηση της, του γενικού αποκλεισμού και της φτώχειας, θα πρέπει και πάλι να, όλα αυτά να μνημονευθούν ρητός ως πολιτική προτεραιότητα. Ακριβώς όπως κάναμε και στο γενικό τμήμα του προϋπολογισμού. Να επομένως, γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι τόσο δόκιμο, δεν είναι τόσο σωστό, παρά την ανεργία και την, ε, και την κρίση, να κάνουμε σε αυτά τα σημεία περικοπή. Τώρα λέμε μετά παραπέρα για το Δάφνη, για το, το πρόγραμμα κατά βίας που πλήσει ανήλικους και γυναίκες. Θα πρέπει και εδώ να υπάρξει μια παραγράφος που σαφώς να αναφέρεται στο θέμα και ρητός. Τώρα, σου φρατη κατηγορία 3β. Και εδώ δεν μας αρέσουν καθόλου οι περικοπές της Επιτροπής, γιατί το 2013 πρόκειται να είναι το έτος του Ευρωπαίου πολίτη και τελευταίο εκεί που αναφέρεται εις όλα τα εξωτερικά μέσα πολιτικής θα πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι όσον αφορά τα κεφάλαια τα οποία αρνούμεθα. Γιατί είδατε τι έγινε με την ε, Αραβική Άνοιξη. Είδατε τι έγινε με το μέσο το προενταξιακό, το Ταμείο σταθερότητας. Όλα αυτά χρειάζονται και χρειάστηκαν επαρκή προοικοδότηση. Αυτά ήταν κάποιες μικρές μικρές πινελιές διορθωτικές διότι καταρχήν μας στο δύο μήκος και με τον κύριο Λαβή όπως σας είπα σας ευχαριστώ πάρα πολύ λέει ο πρώτος και δίνω τώρα στον κύριο Άλβορο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν έχω πάρα πολλά να πω. Έκανε κάθε προσπάθεια ο εισηγητής και αυτό φαίνεται στην ε, έκθεση να συμπεριλάβει όλες τις ε, θέσεις όλων των ομάδων. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνεργασία, ιδιαίτερα χαίρομαι για το ότι δίνεται βάρος σε τομείς σημαντικούς για εμάς, ειδικά σε καιρούς κρίσης δηλαδή να μεταφραστεί πραγματικά σε πράξη η επιθυμία σε καιρούς κρίσης να έχουμε περισσότερες επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, ανατολισμό στόχους του 2020 ε, και βεβαίως ε, έφυξε και το ζήτημα των ε, υπολείπων που έχουν απομείνει σε διάφορους λογαριασμούς ο εισηγητής. Οπότε έχουμε έναν θα πρέπει να έχουμε έναν έξυπνο λογαριασμό, να δούμε να μειωθούν αυτά τα ποσά, τα αδιάθετα υπόλοιπα σε μελλοντικού ε, προϋπολογισμούς. Γιατί έτσι μετά δημιουργούνται χήμερες και προσπαθούν τα κράτη-μέλη να κρατήσουν με τρόπο τεχνητό χαμηλά τον προϋπολογισμό. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Εμείς δεν είμαστε απολύτω σίγουροι για το εάν η φιλόδοξη πρόταση της Κομισιόν ε, για μια αύξηση εδώ πέρα κατά 6% ε, είναι ουσιαστική και αν θα μπορούσαμε να έχουμε αποτελεσματικότερη χρήση των κονδυλίων. Συνολικά λοιπόν θεωρώ πως ε, ο εισηγητής ε, συμπεριέλαβε τις απόψεις της δικής μας ομάδας και είναι σημαντικό αυτό για το μέλλον και το μέλλον της Ευρώπης. Έχω ακόμη μια ε, σκέψη που θα ήθελα να συμπεριλάβω. Σήμερα είδαμε πόσο συναρπαστική μπορεί να είναι η ψηφοφορία για την απαλλαγή των αποκεντρωμένων υπηρεσιών και αναρωτιέται κανείς το εάν η ποικιλομορφία αυτή είναι πραγματικά τόσο απαραίτητη. π.χ. βλέπω εδώ πέρα ρίχνω μια ματιά πως έχουμε και υπηρεσία και ίδρυμα που ασχολείται με ζητήματα εκπαίδευση. Δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε λοιπόν τέτοιες ε, διπλές δομέ. Αυτά ω υποσημείωση ε, επί της αρχής να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο. Νομίζω πως είναι μια καλή και ισορροπημένη αρχή. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για τους αποκεντρωμένους φορείς. Όταν είμαστε σε μια κατάσταση όπως η σημαίνει, στη χώρα μου δημιουργείται μια πρόσθετη αποκεντρωμένη αρχή για να ορθολογικοποιήσει αυτές που υπάρχει. Ο κύριος Άλβαρο. Ε, κύριος Άλβαρο θα ήθελε... Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Χάουκ. Κύριε Άλβαρο. Εγώ έχω ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα. Νομίζω ότι κάνει πολύ ζέστη εδώ πέρα. Πρέπει να έχουμε ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ο οργανισμός μου δεν λειτουργεί κανονικά. Η Μόνικα δεν είναι στην αίθουσα. Δεν θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Έχετε το λόγο Ιούτα και και ο Αλεξάνδρου θέλει να συνεχίσετε. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να πω πως αυτό το οποίο έχει γράψει ο Τζοβάνι πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Ανασένει ευρωπαϊκό πνεύμα αυτός ο άνθρωπος και αυτό βεβαίως ε, δεν μπορεί παρά να μας ικανοποιεί. Επεξεργάστηκε αυτό το οποίο ξεκινήσαμε το 2010 και λέγαμε πως πραγματικά θέλουμε να εφαρμόσουμε και να επιτύχουμε τους στόχους στρατηγικής του 2020 μέχρι το 2020. Δεν τα άφησε για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Είπε τώρα το 2013 πρέπει για αυτούς τους στόχους να κάνουμε κάτι. Και το έκανε πάρα πολύ καλά. Και δεν έχω κανένα παράπονο. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι αναφέρθηκαν οι αποκεντρωμένες ε, υπηρεσίες και ανέφερε και τις δυσκολίες ε, όταν ε, δηλαδή κόβουμε συνεχώς τους προϋπολογισμούς τους γιατί μία μέρα πλέον δεν θα αξίζουν τίποτα. Αλλά το έχω πει εγώ εδώ και καιρό. Γιατί πράγματι σωστό είναι όταν λέμε πως θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να έχουμε ε, κάποια αποτελεσματικότητα. Ναι, αλλά πρέπει να πείσουμε και το Συμβούλιο να συζητήσει αυτά τα πράγματα μαζί μας, αλλά αυτή δεν είναι καν σε θέση να πάνε στην ε, Διοργανική Επιτροπή Συνεργασίας για αυτά τα οποία ήδη έχουμε συμφωνήσει. Το Συμβούλιο, κάποιος το είπε το πρωί, είναι μονίμως σε μια κατάσταση όπου δεν μπορεί, δεν, δεν είναι πλέον ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο και δεν ξέρω δηλαδή πώς μπορούμε να συνομιλήσουμε μαζί τους. Και άλλοι την είχαν την ιδέα. Θεωρώ πως η Ολομέλεια, ε, το, πάντων το αποφάσισε η Ολομέλεια, μπορεί να μου άρεσε, ψήφισε ε, να κλείσει, να συγχωνευτεί ε, η υπηρεσία ισότητας με την υπηρεσία στη Βιέννη. Δεν έχει ούτε μία σχέση. Αλλά τέλο πάντων τι να κάνουμε τώρα είναι τα χέρια μα δεμένα. Το πρώτο είναι αυτό. Ähm, να πω κάτι τώρα για το ψαλίδισμα του προπολογισμού και αυτά τα οποία μας ε, πρότεινε η Κομοσιόν. Επειδή είμαι εισηγήτρια για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, είδα τα νούμερα για το 2013, το, το live. Δεν είμαι μόνο για την επόμενη. Βεβαίω είμαι εισηγήτρια για την επόμενη προγραμματική περίοδο, αλλά πρέπει να ρίξουμε μια ματιά και στο τι γίνεται τώρα. Και πρέπει, βλέπουμε εκεί πέρα, πως η Κομισιόν έχει μια προσέγγιση για το 2013 η οποία είναι κάτω από αυτό το οποίο αποφασίσαμε δια νόμου από κοινού με το Συμβούλιο. Δεν γίνεται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω καν νομικά πώς γίνεται πώς επιτρέπεται. Αλλά ακόμα και αν δεσμεύσουμε και εξοδέψουμε όλα τα λεφτά τα οποία εγγράφονται εδώ πέρα, είμαστε κάτω από αυτά τα οποία έχουμε δεσμευτεί μαζί με το Συμβούλιο. Και συνεχίζεται αυτό ο Τζοβάνι μόλις είπε για το μέσο της αλλά νομίζω πως θα θυμούνται όλοι οι συνάδελφοι πως, ε, ξέρω εγώ πριν από τρεις-τέσσερις εβδομάδες πότε ήταν, ο Μπαρόζο μαζί με τον Μπαν Κιμούν, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, είπανε ενέργεια για όλους. Και είπε 50 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό μας. Ε, πού θα τα βρει. DCI ε, βεβαίως, από πού αλλού αναδιάταξη μέσων εντός του DCI. Οπότε πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά τον προπολογισμό και να μας εξηγήσει και η Κομισιόν πώς έχει κάνει τους υπολογισμούς της. Και πιστεύει ότι βγαίνει. Αλλά κάτι άλλο που με ενδιαφέρει Τζοβάνι. Στην αρχική σου δήλωση μίλησες για τη χτεσινή εκδήλωση στη χθεσινή εκδήλωση. Μίλησε με την Κομισιόν για τις πληρωμές και εκεί πέρα πληροφορήθηκε πως η Κομισιόν έχει αξιολογήσει πολιτικά τις πληρωμές. Ε, έχει κάνει μια πολιτική στάθμιση των πληρωμών. Για εξήγησε το μου αυτό. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Τι πάει να πει πολιτική στάθμιση των πληρωμών. Merci, Francesca Oui, merci. Euh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να πω πως ε, πραγματικά στηρίζουμε την έκθεση και ευχαριστούμε τον ε, εισηγητή. Ε, βεβαίως θα καταθέσουμε κάποιες ε, έτσι, τροπολογίες για το πρασίνισμα. Θεωρώ πως στην κρίση αυτή πρέπει να φροντίσουμε να βγούμε καλύτεροι από την κρίση από ό,τι μπήκαμε, με οικονομίες πιο ανταγωνιστικές και αποτελεσματικές, ειδικά όσον αφορά τη χρήση πόρων και ενέργειες. Θα καταθέσουμε στροπολογίες, αυτό το ξέρετε, αλλά σε καιρό κρίσης αυτό είναι βασικό. Και είναι σημαντικό, όπως τονίσατε, να υπερασπιστούμε τα επίπεδα που ζήτησε η Κομισιόν και θα είναι δύσκολο αυτό από πλευράς επικοινωνίας, αλλά όπως είπε και η Γιούτα, πρέπει να είμαστε ισχυροί ως προς αυτό και υπέρ της Ευρώπης δεν μπορεί να λέμε πώ χρειαζόμαστε το ένα και το άλλο και μετά να κόβουμε όλου του προπολογισμού. Πρέπει να τα υπερασπιστούμε αυτά από κοινού. Και θεωρούν πω είναι καλή ιδέα να ορίσουμε αρνητικέ προτεραιότητε Υπό αυτή την έννοια. Ναι, αυτό είναι κάτι θαραλέο και το στηρίζουμε. Από την άλλη, βλέπουμε πως οι φόβοι μας επαληθεύονται όταν μιλάμε για τη χρηματοδότηση του Twitter. Δεν χαιρόμαστε, αλλά είχαμε δίκιο. Είναι θλιβερό γιατί βλέπουμε πως παίρνουν λεφτά από άλλα μέρη του προγράμματος πλαισίου 7 και είναι λάθος αυτό. Στον τίτλο 4 μπορώ να πω πως θα συμφωνήσω με αυτό το οποίο είπαν άλλοι για τις περικοπές στο DCI, για τη σταθερότητα. Δεν είναι σαφές γιατί κόβουμε εκεί πέρα γιατί ήταν σαφές νομίζω πως ε, πολλές από τις υποσχέσεις που έχει κάνει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης κάπως πρέπει να πληρωθούν. Και βλέπουμε πως κόβονται τώρα. Ειδικά, αυτό είναι αρνητικό, ειδικά γνωρίζοντας πως ε, για τα επόμενα 7 χρόνια θα αποτελέσει αφετηρία ο προπολογισμό του 2013. Και είναι θλιβερό να κόβεται άρα ο προπολογισμό του 13% κάτι το οποίο θα επηρεάσει το επόμενο επταετέ πλαίσιο. Και κάτι άλλο που αναφέρατε ήδη όσον αφορά την νεολαία σε κίνηση και την διαβίου μάθηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά, ειδικά όταν οι πολίτες απομακρύνονται από την Ευρώπη. Υπάρχουν κάποια προγράμματα τουλάχιστον που επηρεάζουν άμεσα τις ζωές των ανθρώπων και πρέπει να συνεχιστούν και να αυξηθούν οι δυνατόν. Το αναφέρατε αυτό. Και συμφωνούμε. Θα καταθέσουμε λοιπόν κάποιες τροπολογίες όπως είπα. Στα υπόλοιπα συμφωνούμε με τους περισσότερους ομιλητές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σταυρακάκης. Thank you very much, Mr. Chair. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να και τον εισηγητή, τον κύριο Λαβία θα ήθελα να λάβω το λόγο σαν εισηγητής για τα θέματα του προϋπολογισμού στην Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων. Πρέπει να δούμε τον προϋπολογισμό μέσα στα πλαίσια της, ε, της οικονομικής κρίσης και των περιορισμών που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Σε όλα τα κράτη της Ευρώπης γίνονται προσπάθειες δημοσιονομικής παγιοποίησης και μέτρα λιτότητος. Αλλά είναι σημαντικής, ε, μεγάλης σημασίας να αντισταθμίσουμε αυτή την εδραίωση με επενδύσεις οι οποίες θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και οι οποίες θα επιτύχουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα στα πλαίσια αυτά η πολιτική συνοχής έχει καταδείξει την προστιθέμενη της αξία ως εργαλείο το οποίο οδηγεί σε ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης για να αντιμετωπίσει και τις ανάγκες επενδύσεως των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, οι περιφέρειες μπορούν να συμμετάσχουν στην συνολική ανακάμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ξέρουμε, η βελτίωση της εφαρμογής των περισσότερων προγραμμάτων στην κατηγορία 1β οδήγησε στο τέλος του 2011 σε, πολύ, σε πολλές πληρωμές οι οποίες επίκυνται που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με αυξημένε πιστώσει υποχρεώσεων το 2013. Έχουμε ανησυχίε ότι όλα αυτά μπορεί να επιδεινωθούν και το 2013 γιατί η κατηγορία 1β, η εκταμείευση στην κατηγορία 1β θα κινδυνεύει να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Για το λόγο αυτό, στη γνωμοδότησή μου της Επιτροπής ε, Περιφερειακών Θεμάτων, ζητώ από το Συμβουλίο να αναλύσει τα στοιχεία αυτά μαζί με την Κομισιόν ώστε να μην τεθεί ένα αμφιβόλο η εφαρμογή των κονδυλίων αυτών το 2013. Υπάρχουν πολλοί, πολλές περιοχές με καλά προγράμματα που βρίσκονται σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή. Ζητώ επίσης από την Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων μαζί με την Κομισιόν και το Συμβούλιο να εξετάσει ενδελεχώς τις ανάγκες πληρωμών στην κατηγορία 1β που βασίζονται και στις προβλέψεις των κρατών μελών και που έχουν αποτελέσει και τη βάση για το σχέδιο προϋπολογισμού. Κλείνω να σας πω ότι επί τη βάση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2013 που παρουσίασε ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι στην Επιτροπή μας θεωρώ ότι η αύξηση που προβλέπεται στο σημείο στην κατηγορία 1β είναι πολύ καλό σημείο έναρξης των διαπραγματεύσεων για το 2013 αλλά δεν θεωρώ ότι θα είναι επαρκής δυστυχώς. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ο Σαλβαδόρ Γαρίγα που λέγεται τώρα Νιένσκι. Ναι, ναι, ακριβώς. Λέει ο μιλητής. Ναι, εγώ σας μιλώ τώρα ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, γιατί θα πρέπει να ευχαριστήσω τον Τζοβάνι Λαβία για το σχέδιο έκθεσης, το οποίο αφορά τη διαπραγματευτική εντολή για τον προϋπολογισμό και είμαστε στο ίδιο μήκο κύματος μετά όσα είπε εκείνος. Όμως θα πρέπει σε σχέση με κάποιες επιφυλάξεις που στη συζήτηση ανεφύσαν, να σας πω ότι το σχέδιο προπολογισμού το οποίο λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να κατευθυνθεί προς δύο δύσκολα θέματα ε, το ότι χρειάζεται να καλύψουμε τις τις δημοσιονομικές εντάσεις, την κρίση, την δημοσιονομική λιτότητα, αλλά και δεύτερον να ενισχύσουμε τις πιστός πληρωμών, ούτως ώστε να παρακάμψουμε προβλήματα σαν τα σημερινά, εκεί όπου δηλαδή έχουν φρενάρει οι πληρωμές. κ. Σκοτσμάν, επίσης, ο οποίος ακάματα εργάζεται προ αυτή την κατεύθυνση και θεωρώ ότι κάποιε από τις τροπολογίες είναι πάρα πολύ σωστέ, 15 κράτη-μέλη ε, είδαν να παγώνουν οι πόρε τους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και βέβαια με την κρίση τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί με τίποτα να κάνει αυτό το οποίο οφείλει λόγω του αυτών των προβλημάτων στις πληρωμές. 15 είπαμε ε, κράτη-μέλη έχουν πρόβλημα με το Γενικό Ταμείο και άλλα 9 με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφέρειας Ανάπτυξης οπότε θα πρέπει ο κύριος ε, Λαδία να παλέψει κατά των χαμηλών αριθμών ανάπτυξης και που θα πρέπει να, να, να διορθώσουμε και των πιστώσεων πληρωμών που θα πρέπει να ανεβούν. Βεβαίως, οι πιστώσεις ή συμβαστικού χαρακτήρα θα πρέπει και αυτές να καλυφθούν. Και αυτές οι πιστώσεις υποχρεώσεων θα πρέπει στο, στη χρήση του 2013 να είναι τέτοιες που να αντιστοιχούν με την ανάπτυξη που θέλουμε για να δημιουργήσουμε κάποια απασχόληση στην Ευρώπη. Γι' αυτό αγαπητοί συνάδελφοι, Όσον αφορά την εντολή του προπολογισμού που θα ξεκινήσει τη διαδρομή του το Σεπτέμβριο, θα πρέπει να μην αποκλίνουμε από την πορεία, από τη ρότα του να κάνουμε κάτι για τις πληρωμές. Επομένως, 100% να υποστηρίξουμε το κείμενο της προτάσεις, δηλαδή για τις πληρωμές, γιατί η οικονομική ανάπτυξη ε, ε, ε λόγω της λιτότητας του 2013 θα έχει βάση της, θα έχει κινητήρια δύναμη με αυτές τις πιστώσεις πληρωμών. Να δούμε τι θα κάνει το, η Κομισιόν, τι θα κάνει το Συμβούλιο, προς τους οποίους εμείς θα, κατεβάσουμε μια άλλη ανεξάρτητη πολιτική πρόταση για τις πληρωμές για τη χρήση 13 και οπότε ως προς αυτό θα πρέπει όλο το πολιτικό βάσμα του Κοινοβουλίου να στηρίξει τις προτάσεις δηλαδή ε. ο Πρόεδρος. Σαρβαντό, ευχαριστούμε. Ο κύριο Κοτμάνης έχει το λόγο. Για άλλη μια φορά, κύριε Κοτμάνης, έχετε ετοιμάσει αυτό τα πινακάκια. He saved also my time. Uh, for that reason I will not repeat what... Τα είπε ο Σαλβαντόρ, με έσωσε και με κάλυψε, αλλά εγώ θα πω άλλα. Σήμερα είδαμε τις προτάσεις για τη μεταφορά των πιστώσεων Μιλάμε για 350 εκατομμύρια για αυτό το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της οικονομίας. Και πολύ σωστά ετέθη το ερώτημα. Τι έγινε, τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα, θα προωθηθούν ή όχι. Και θυμάμαι ότι όταν αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε δεν ήμουν ευρωβουλευτής αλλά ήμουν Πρωθυπουργός και πολύ χάρηκα και ξαφνικά εκεί από ε, τη μικρή μας πατρίδα είδα, είχαμε 72 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα, θα, θα, θα ερχόντουσαν στο μάνα εξ ουρανού και όμως το, πρόγραμμα, το πρόβλημα ήταν ότι καταλήγουμε τώρα να, να, μας, να έχουν παγώσει 5 δις και ένα δις ακόμα πιστιστή βοήθεια όμως υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει σπάνιες για τους πόρους. Τι θα κάνουμε. Δεν νομίζω ότι τα η Κομισιόν έγινε ψηφοφορία και εμείς ψηφίσαμε προς αυτή την κατεύθυνση για αυτούς τους πόρους. Όχι, δεν το αποφάσισε μόνη της η Κομισιόν. Όλοι έχουμε κοινή ευθύνη. Αντιδράσαμε γρήγορα όσον αφορά την κρίση, αλλά για την ενεργειακή υποδομή μιλάμε για μεγάλη διαδρομή. Υπάρχουν θέματα ε, απαλωτριώσεων, είναι θέματα δικτύων κλπ. Για να δούμε. Θα πρέπει κάποιος να μας πει με ακρίβεια τι γίνεται. Εάν κάποιος τα διρεαλιστικά θα διαπιστώσει ότι αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να απορροφηθούν ή θα απορροφηθούν σε 50 χρόνια για να γίνει ο σωστός προγραμματισμός. Θα πρέπει με θάρρος να πει κάποιος αγαθές και επενετές προθέσεις σας, αλλά από πλευράς πραγματικότητας δεν γίνονται αυτά. Να έχουμε ένα μικρό αποθεματικό για να καλύψουμε τις ανάγκες τα είδα, τα βλέπετε σε αυτό το πινακάκι που σας μίλησα. Δεν είναι θέμα οικονομικών ελέγχων. Είναι θέμα ρευστότητας. Τα έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 5-6 δις είναι η μία προωθηθήσεις πιστώσεις. Τι να κάνουμε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, κόβουμε λεφτά από ένα, τα δίνουμε σε άλλον, αλλά είναι ρεαλιστικό να ποντάρουμε σε κάποιο αποθεματικό, γιατί το πρόβλημα είναι ότι το πρόβλημα της πληρωμές θα έχει τις εξής συνέπειες. Πρώτα πρώτα, πρώτα, πρώτα για την ανέψη της πέθρου, δεύτερον για τη συνοχή και για την έρευνα και ανάπτυξη. Και βέβαια τα πράγματα γίνουν πιο μπερδεμένα γιατί δεν αποφασίζουν οι τεχνοκράτες της Ένωσης αλλά επιστήμονες για το ποια προγράμματα και project θα εγκριθούν. Άρα ούτε εκεί είναι προβλέψιμα τα πράγματα. Και το ερώτημα που αναδύεται είναι το εξή. Εάν θεωρηθεί ότι δεν έχουμε αποθεματικό, τι θα γίνει. Έχουμε αυτό το 6,8% για το οποίο κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι θα κάνει το Συμβούλιο. Τι θέλουν να παρελκύσουν την κατάσταση για να πάμε στην κατάσταση που επικρατούσε το 2012 από ήταν τα πράγματα στι 11. Θα πρέπει. Εάν έχουμε 6,8 και όχι περισσότερο, να δούμε ποιοι προτίθενται να βοηθήσουν για αυτές τις πληρωμές και, τι, και να κάνουν κάτι για αυτά τα οποία δεν θα εκταμιευθούν ή δεν θα απορροφηθούν φέτος και θα μεταφερθούν για το μέλλον. Δεν υπάρχει άλλο, άλλη λύση, άλλος τρόπος. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πόσες χώρες θα καλυφθούν. Ε, φτά. Λέμε εδώ πέρα και πολλέ φορέ για ειδική πλειοψηφία, ενισχυμένη πλειοψηφία, αλλά αυτά δεν ισχύουν για το Συμβούλιο. Επομένω, α μα πει κάποιο υπεύθυνα τι δυνατότητε υπάρχουν για μια λύση από πλευρά αποθεματικού και δεύτερον τι γίνεται από πλευρά ρευστότητα. Κάποτε η Κομισιόν είχε θέσει ένα αυστηρόχρονο διάγραμμα για δύο από αυτά τα ταμεία και είχε πει εάν δεν κάνετε ακόμα και η Γερμανία αυτό που πρέπει δεν θα πάρετε τα λεφτά που θα τα χάσετε. Ας έρθει η κυρία Χιμπνερ για να μας πει τι έγινε με αυτή την καταληκτική ημερομηνία. Κάποιε κάποιες χώρες πήγανε παραπέρα, πήγαμε στο 10, πήγαμε στο 11. Και αν δείτε τις πληρωμές από πάσης απόψεις από, από, από παντού θα δείτε ότι έχουμε ένα σωρό χρήματα και αυτοί οι πόροι δεν θα ξέρουμε ποιος θα τους, ποιος πού θα πάνε. Άρα, ή κάποια χρήματα δεν θα εκταμιευθούν Έχουμε τη διαγράμμιση του Πέτρου, έχουμε τη συνοχή, έρευνα, ανάπτυξη. Λοιπόν, δεν πρόκειται αυτά να εκτενευτούν, διότι και κάποιε χώρε δεν ετήρησαν τι υποχρεώσει του με το τεθέν χρονοδιάγραμμα. Ή αυτό, ή να δούμε ε, ρεαλιστικά. Γίνεται από κάποιο αποθεματικό να πάρουμε κάποια χρήματα για, για κάποιες ε, αποκρισταλωμένες, για κάποιες σύνομες πληρωμές. Κάποιε χώρε έχουν καθυστερήσει κατά, κατά Και δεν μιλάω και για, για αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά ταμεία. Μιλάω για κάποια άλλα δευτερεύοντα, τα πούμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που σα λέω τώρα, διότι έχει να κάνει με τι αποφάσει και προτάσει Λαβία. Και αυτά τα ζήτησε και, το, και, και ομάδα εργασία για το, για το πλαίσιο. Να δούμε επομένω πόσο και αν μπορούμε να αναβάλουμε και να μεταφέρουμε για το μέλλον. Δυστυχώς όλα αυτά όμως αλληλοσυνδέονται. Και άρα με πολιτικές αποφάσεις το να κρατά κανείς τις πληρωμές σύμφωνοι γίνονται αυτά αλλά τι θα γίνει μετά από 7 χρόνια με το πολιετές ε, πλαίσιο εκεί πια είναι θέμα συνθήκης, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Γι' αυτό σας λέω, είναι πάρα πολύ σωστές οι προτάσεις Λαβία, αλλά το ερώτημα είναι τι θα γίνει. Δεν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να, να, να μαλώσουμε κανένα. Δεν θα υπάρξει αντιπαράθεση, αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά τα έκτακτα μέτρα για την κρίση. Κανείς δεν μπορεί να μας κατηχωρήσει. Κανείς δεν μας κατηγορήσει. Και κανείς δεν μπορεί επίσης να πει, εάν δεν έλαβαν αυτά τα μέτρα, τι θα είχε συμβεί. Όλοι όσοι ήταν σε, σε κυβέρνηση, στο τιμόνι μιας χώρας το 8, τώρα όλοι έχουν πέσει εκτός από τη Μέρκελ και το Τούσκης. Άρα, τι γίνεται με την πειθαρχία, τι γίνεται με τα αποθεματικά, τι γίνεται με τη ρευστότητα, για να δούμε για αυτή την εφταετία του πολιετούς πλαισίου τι θα κάνουμε. Και συγγνώμη μακρηγόρησα. Merci, mon cher collègue, pour cette... Euh, Ευχαριστώ αγαπητέ <clears throat> συνάδελφοι για αυτή τη λαμπρή ανάλυση και για τη συνολική παρουσίαση που μας κάνετε. Κύριε Σιγητά, τι συμπεράσματα ανα, έχετε ανακτήσει από όλα αυτά τα οποία έχουν ελεγχθεί. Μετά από αυτά που είπε ο κύριος Άλβαρο και εγώ, και εγώ ένιωθα να ανεβαίνει η θερμοκρασία και να υδρώνω, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό για ένα εισηγητή, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα το καλοκαίρι και δεν έχουμε τελειώσει με τις προτάσεις των ε, συναδέλφων. Και, και άλλοι νιώθουν ότι έχει ζέστη σε αυτή την αίθουσα, Επομένω χαίρομαι γιατί δείχνει ότι δεν είμαι εγώ μονάχα που νιώθω κάποιο εκνευρισμό. Σε σχέση με αυτά τώρα που είπαν οι διάφοροι συνάδελφοι, είναι φανερό ότι από τις διάφορες παρεμβάσεις των πολιτικών ομάδων μπορώ να διαπιστώσω ότι υπάρχει γενική συμφωνία με την γενική πλατφόρμα με τα βασικά στοιχεία λοιπόν της εντολής του τριγωνικού διαλόγου. Προφανώς θα υπάρξουν επιμέρους διαφοροποίησεις των πολιτικών ομάδων επί τη βάση των δικών τους προτεραιοτήτων. για να καταδείξουν και ορισμένε διαφορές που έχουν. Όταν βλέπω παραγωγούς χάρη τους πράσινους, καταλαβαίνω ότι θα προτείνουν για το σχέδιο ΙΤΕΡΤ και φυσικά θα είναι οι προτάσεις και οι τροπολογίες αντίστοιχες με αυτές που έχουμε δει και τα προηγούμενα έτη. Θέλω να πω όμως κάτι σε σχέση με αυτό που ελέγχθη για ορισμένε συγκεκριμένες γραμμές του προϋπολογισμού για την κατηγορία 4 και άλλες κατηγορίες όπου κάποιες από τις περικοπές που έχουν γίνει στην πρόταση της Κομισιόν βλέπουμε ότι συσχετίζονται άμεσα με την έλλειψη επαρκούς απορρόφηση αυτών των γραμμών του προπολογισμού τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Κομισιόν έχει ήδη <clears throat> διατυπώσει αυτές τις αναθεωρημένες προτάσεις, γιατί αυτές οι γραμμές της, ε, του προϋπολογισμού δεν ε, έχουν δείξει την ικανότητα πλήρους εκταμίευσης. Γι' αυτά που είπε η Ιούτα, μίλησε για μια πολιτική στάθμιση των πληρωμών. Η Κομισιόν έχει διατυπώσει κάποιες προβλέψεις λαμβάνοντας πάντα υπόψη το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει μεγάλη χρησιμοποίηση στην πολιτική συνοχής. Κάποιο τμήμα των πόρων λοιπόν ούτως ή άλλως δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη-μέλη. Αλλά η πρόταση η αρχική των ε, επιτρόπων ήταν πιο υψηλή σε σχέση με τις πιστώσεις πληρωμών και στη συνέχεια αναθεωρήθηκε από την Κομισιόν. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά είναι μια πολιτική εκτίμηση και υπήρξε επομένως μια διόρθωση για τα θέματα αυτά. Είναι γεγονός ότι το θέμα των πιστώσεων πληρωμών που αναφέρθηκε σχεδόν από όλους θα είναι και το κεντρικό θέμα της συζήτησής μας, όπως έλεγε και ο κύριος Γκαρίγκα. Και είναι το θέμα για το οποίο εμείς θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτά που είπε ο κύριος Κοντμάνης και ο πίνακας τον οποίο παρουσίασε, προφανώς θέτουν ανάγλυφα ένα συγκεκριμένο ζήτημα για το οποίο θα πρέπει μέσα σε αυτό το έτος να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες οι οποίες θα προκύψουν. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του επίπεδου εκταμίευσης και ο διορθωτικός προϋπολογισμός που θα προκύψει στο τέλος του έτους επί τη βάση των προβλέψεων που θα υποβάλουν τα κάτι μελη μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλα αυτά θα μας δώσουν ορισμένε συγκεκριμένε ενδείξεις για το αν για του χρόνου θα πρέπει να παραμείνουμε στην ίδια κατάσταση που είμαστε φέτος ή σε χειρότερη ή σε βέλτια κατάσταση. Επομένως όλη η συζήτηση για τις πιστώσεις πληρωμών θα πρέπει να συνδεθεί με τον απολογισμό του 2012. Γιατί εάν δεν μπορέσουμε να καλύψουμε τις πληρωμές του 2012 και πρέπει να μεταφερθούν κάποιες από αυτές το 2013, θα έχουμε μια πλημμυρίδα, ένα τσουνάμι, μια αυξανόμενη ποσότητα κονδυλίων και θα βρεθούμε λοιπόν σε μια πολύ δύσκολη θέση. Θα έχουμε λοιπόν το τσουνάμι το οποίο θα μπει στο λιμάνι και θα καταστρέψει πολλά πράγματα. Κλείνω με το εξή σημείο. Αναφερθήκατε για μια ευφυά διαχείριση του προϋπολογισμού. Ναι. Αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με μεγάλη προσοχή. Ο καθένας αγαπάει τα πράγματα που κάνει φυσικά, αλλά θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να δούμε μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, στην κάθε επιτροπή ο καθένας, που μπορούμε να περικόψουμε τις δαπάνες όχι μονάχα γιατί οι γραμμές του προϋπολογισμού δεν είχαν την επαρκή εκταμίευση για τα θέματα αυτά, αλλά και επειδή ίσως μπορεί να θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα για την ανάπτυξη, για την, ε, τον ανταγωνισμό, την ε, απασχόληση για ορισμένε πρωτοβουλίε μπορούν να είναι μεγαλύτερε οι δυνατότητε για ορισμένου τομεί και μικρότεροι για άλλου. Γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με ευφυα του πόρου που θα έχουμε στη διάθεσή μα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ κύριε Σίγητα. Σας ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω ότι σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτή η υποθεσμία τροπολογιών 31 Μαΐου το μεσημέρι θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Προϋπορεσμό στις 20 Ιουνίου και στην Ολομέλεια ως ήθιστε τον Ιούλιο. Σας ευχαριστώ κύριε εισηγητά. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε μετά από όλα αυτά εντάχει στο σημείο 5 την διαπραγμάτευση για, τους, για τις πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές. Μα δεν είναι εδώ οι συγητές. Α, εδώ, συγγνώμη, είναι νέο. Ναι, ο Ήβαλο Ελά είναι παρόν, συγγνώμη. Απλώς για καλύτερη πληροφόρηση των μελών και του κοινού που μας παρακολουθεί να κάνω μια ενημέρωση για τις τελευταίες ε, συνομιλίες που κάναμε χθε με τη δανική Προεδρία από τη μία πλευρά, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου από την άλλη μεριά και την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Προεπολογισμών Και επίσης σήμερα πάλι τη συζήτηση που έγινε στην ομάδα επαφής με την παρουσία του Προέδρου Σούλτς. Έχουμε πολλές φορές και ιδίως χθες τονίσει στη Δανική Προεδρία ότι σε ό,τι αφορά εμάς την ε, Επιτροπή Προϋπολογισμών που έχουμε σαν ομόλογο τον κύριο Βάμεν για Υπουργό Εξωτερικών Επομένως για τις ε, γενικές υποθέσεις και αντίστοιχα έχουμε εκφράσει τις ανησυχίες μας για τα λεγόμενα κοιτία διαπραγμάτευσης Επομένως τα έγγραφα τα οποία θα μας δώσει το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, μάλλον θα δοθούν πρώτα στο, Συμβούλιο Γενικών, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου και σε σχέση με την στάση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα θέματα αυτά. Γιατί η θέση μας είναι ότι δεν πρέπει να καθορίσει πρόωρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα αριθμητικά ποσά ούτε για το γενικό ποσό, το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, ούτε για τους διάφορους τομείς και δεν πρέπει να, καταλα... να πάρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λεπτομεριακές αποφάσεις για θέματα τα οποία υπόκεινται στην συναπόφαση. Πρέπει να διατηρήσουμε λοιπόν και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου και τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης του ίδιου του Κοινοβουλίου σε μια στιγμή που τα θέματα αυτά αρχίζουν να συζητούνται περισσότερο σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όχι σε επίπεδο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, όπως ήθιστε. Ελπίζω ότι αυτό το μήνυμα έγινε αποδεκτό και για να είμαι σίγουρος ότι η Ιδανική Προεδρία θα το λάβει υπόψη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίσης θα λάβει υπόψη το σημείο αυτό, εμείς κινούμεθα προς την κατεύθυνση της έγκρισης μιας, ενός ψηφίσματος στο, στην Ολομέλεια πριν φτάσουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να υπενθυμίσουμε με αυτό το σύντομο, με ένα σύντομο κείμενο, δύο σελίδων το maximum, ποιε είναι οι ουσιαστικέ προτεραιότητε, ποιε είναι οι βασικέ ανησυχίε μα, ποιε είναι οι κόκκινε γραμμέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι διαπραγματεύσει αυτέ. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζουμε είναι πότε θα υποβληθεί στην ε, Ολομέλεια αυτό το ψήφισμα. Θα γίνει αυτό στην επόμενη συνεδρίαση του Μαΐου 2 στο Στρασβούργο ή τον Ιούνιο. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να περάσουμε αυτό το ψήφισμα το Μάιο ή δυνατόν, γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να γίνει και δημόσιο αυτό το ψήφισμα, προτού να περατωθεί το θέμα των κοιτίων διαπραγμάτευσης από το από τους Υπουργούς Γενικών Υποθέσεων. Επομένως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μέσα στα πρακτικά των διαπραγματεύσεων που θα διαβιβαστούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η άλλη επιλογή θα ήταν να εγκριθεί αυτό το ψήφισμα τον Ιούνιο ανάμεσα στις συνεδρίες του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η τελική απόφαση φυσικά θα για αυτά τα θέματα θα ληφθεί από τους πρόεδρους των πολιτικών ομάδων και έχουμε συμφωνήσει ότι σε μια χρονική εποχή όπου δυστυχώς η οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση είναι ιδιαίτερα βεβαρημένη και αλλάζουν τα πράγματα είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Έχουμε τις ανησυχίες για την Ελλάδα, για την Ισπανία, και άλλες χώρες όπου επίσης έχουμε τις πολιτικές αλλαγές στη Γαλλία. Υπάρχει το έκτακτο συμβούλιο το οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που προβλέπεται στις 23 Μαΐου, που είναι η τετάρτη της Ολομέλειάς μας στο Στρασβούργο. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα η συζήτηση αυτή που προέβλεπε να προτείνει ο πρόεδρος Σούλτς σε σχέση με την έγκριση αυτού του ψηφίσματος με παρουσία του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του εκπροσώπου της Δανικής Προεδρίας φυσικά δεν θα μπορέσει να λάβει χώρα γιατί κατά πάσα πιθανότητα οι συνομιλητές μας θα είναι στις Βρυξέλλες στην προετοιμασία ή στη διεξαγωγή του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για τη συγκεκριμένη λοιπόν ημερομηνία δεν έχουμε ακόμα κάποια συμφωνία. Προετοιμάζουμε από την πλευρά της ε, Αντιπροσωπείας της Επιτροπής Προϋπολογισμών ένα προσχέδιο το οποίο θα υποβληθεί για το ψήφισμα αυτό στην ομάδα επαφής και στην σύνοδο των Προέδρων και εν καιρό όλα αυτά θα έρθουν στην Ολομέλεια. Αυτά λοιπόν. Και οι ειδικευμένε και εξειδικευμένε μας επιτροπές θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά για τις επιμέρους πολιτικές. Ήβαλο θέλετε να πείτε κάτι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ένα πράγμα. Εξηγήσατε με λεπτομέρειες το τι συμβαίνει στις ε, διαπραγματεύσεις. Να προσθέσω κάτι ακόμα. Να ξέρουν οι συνάδελφοι πως στην τελευταία συνάντηση, τη χθεσινή συνάντηση μεταξύ πρόεδρου Σούλτς και του Υπουργού του κυρίου Βαμμένη, η Προεδρία της Δανίας άνοιξε μια χαραμάδα για κάποια νούμερα στο, στην απόφαση του Συμβουλίου του Ιουνίου. Βεβαίως αυτό είναι κατά το Κοινοβούλιο γιατί πριν ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις ε, για την πολιτική δεν θέλουμε ε, να δούμε νούμερα βεβαίως. είπε η Προεδρία της Δανίας πως πιθανότατα δεν θα υπάρχουν νούμερα αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς πως δεν αποκλείεται 100% η πιθανότητα από πλευρά Προεδρίας της Δανίας πλέον. Αυτό θα ήθελα να, να προσθέσω εγώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να τελειώσουμε με αυτό το θέμα και να περάσουμε στο βαθμό 6. Φραντσέσκα, συγγνώμη να σας αποσπάσω λίγο από τη συζήτηση με τον διαδοχό σας για να μας ε, παρουσιάσετε το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 3. Ευχαριστώ. Ο προϋπολογισμός ο διορθωτικός υπαριθμών 3 αφορά το πλεόνασμα, το οποίο δεν είναι τόσο μεγάλο όσο ήταν πέρσι. Βεβαίω πέρσι ήταν 4,54 δισεκατομμύρια, φέτος είναι 1,49 δισεκατομμύρια. Το πλεόνασμα είναι αρκετά ισορροπημένο, περισσότερο, υπήρχαν περισσότερα έσοδα, 6,67 δισεκατομμύρια και δαπάνες 728 ε, εκατομμυρίων και 47 εκατομμύρια από τις διακοιμάνσεις ε, της ισοτιμίων. Οπότε συνολικά έχουμε κάποια εξοικονόμηση, ένα μεγαλύτερο εισόδημα το οποίο βεβαίως γίνει ούτω ή άλλω ε, ουδέτερο γιατί θα επιστρέψει στα κράτη-μέλη και θα μειωθούν οι συνεισφορέ τους. Μιλήσαμε για το ότι είναι κατάλληλο να διατηρηθεί αυτό ο μηχανισμός όταν παραπονιόμαστε κάθε μέρα για το ότι δεν έχουμε αρκετές πιστώσεις πληρωμών και πιθανώς αυτό είναι πιο τεχνικό έγγραφο παραπολιτικό και ίσως θα έπρεπε να έχουμε κάποιες εκθέσεις για να μιλήσουμε ίσως πριν από την Ολομέλεια για το πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πιθανώς αυτό το πλεόνασμα με τρόπο διαφορετικό έτσι ώστε να βοηθήσει τον προπολογισμό της κοινότητας και να μην επιστραφεί στα κράτη-μέλη. Οπότε θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και μετά θα μας πει την άποψή του το Συμβούλιο και θα συζητήσουμε μετά την έκθεση στην Επιτροπή και μετά στην Ολομέλεια βεβαίω. Σας ευχαριστώ. Περνάμε σημείο 7 καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Aider. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα ήθελα σήμερα, πέραν του να κάνω την εισήγηση για αυτή την έκθεση που ακόμα είναι υποδιαμόρφωση, είναι το να ανοιχνεύσω λίγο τις απόψεις εδώ των συναδέλφων για να δω πού το πάνε. Μια που Βέβαια έτσι και αλλιώ τα πράγματα. Το πρόγραμμά μα κάπω φορτωμένο, μια που έχουμε τώρα τη Να σα πω τέλο πάντων δύο λόγια, να σα πω δύο-τρία δύο, στοιχεία τα οποία ίσω ενδιαφέρουν. Πρώτα-πρώτα το χρονοδιάγραμμα. Ε, αυτό το οποίο θα ήθελα είναι το σχέδιο κειμένου να σα το προσθέσω κατά τα τέλη Μαΐου ούτω ώστε να υπάρξει χρόνο μετάφραση σε όλε τι γλώσσε και μετά στι 21 Ιουνίου, όπου εκπνέει η σχετική προθεσμία, να έχουμε τι ε, τροπολογίε και να κάνουμε την ε, ψηφοφορία στην υποτροπή μα καταρχήν τον Ιούλιο. Βεβαίω ε, έχουμε τι γνωτήσει Ήτρε, Ρέτζι και Κοκομπού που πάνε προς την ίδια κατεύθυνση στόχος για αυτής της έκθεσης είναι ακριβώς το να έχουμε μια συγκεκριμένη αλλά και ε, να καλύπτει πολλά γενικά πράγματα η Επιτροπή αυτή για όχι να αναλύσουμε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, να δούμε ποια, ποιο είναι το θεμέλιο, ποια είναι η βάση ε, από την οποία ξεκινάνε και στην οποία στηρίζονται αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα. Έχουμε τέσσερις, ε, τέσσερα κομμάτια. Πρώτα-πρώτα τον ορισμό του τι ορίζεται χρηματοοικονομικό μέσο. Υπάρχουν πολλές απόψεις, είναι τεχνικό αυτό το θέμα Επομένως θα ήταν ε, σωστό να έχουμε μια πρώτη ε, διευκρίνηση για το τι ισχύει για τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Να κάνουμε επίσης μια αξιολόγηση για το πώς λειτουργούν αυτά τα μέσα ε, και πριν την τυρκουάζ εβδομάδα να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με κάποιους ειδικούς εμπειρογνώμονες να μας πούν που βλέπουν τα πλειονεκτήματα, βλέπουν τα μείον αυτών των μέσων ε, να μας πούν πώς μπορούμε να κάνουμε κάποιες διορθώσεις και μετά να κάτσουμε για να αξιολογήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα μέσα αυτά, για το, για το πλαίσιο αυτό 2014-2020 οπότε και κυρίω θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι έχει γίνει κάποιο βήμα προς τα εμπρός να μας παρουσιάσει μία έκθεση η Επιτροπή να ξέρουμε και περισσότερα από όσα είχαμε στα χέρια μας μέχρι τώρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο για τη διαδρομή που θέλω να κάνω και να δω μέχρι πού, μέχρι πότε μπορούμε να φτάσουμε με αυτά τα μέσα, τι τάξεις μεγέθουν αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα, πώς μας εξυπηρετήσουν τον προπολογισμό. Στις συναντήσεις που έχω κάνει μέχρι σήμερα, είπαμε και ξαναείπαμε διάφορα, πολλά θέματα. Αυτά που θα τα συζητήσουμε και εδώ. Πάντως, εγώ θέλω να σταθώ στο ότι αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα για να λειτουργήσουν, για να αποδώσουν, θα πρέπει να έχει προηγηθεί ανάλυση εντελεχής για το πώς έχουν τα πράγματα τι είδου καταλήτες είναι για την αγορά και μετά να τα θέσουμε σε ισχύ και έτσι μετά να αποσπάσουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Θα πρέπει να έχουν πάντως μια εσωτερική συνέπεια, μια εσωτερική συμβατότητα για να πιάσουν τόπο. Αλλά κυρίως θα πρέπει να είναι ευέλικτα, διότι τη σήμερα ημέρα υπάρχουν προβλήματα στην αγορά αλλά από την άλλη μεριά και εμεί θα πρέπει να είμαστε προσαρμοστικοί όσον σχέση με το τι χρειάζεται τώρα. Μια επίκριση η οποία τώρα διατυπώνεται όσον αφορά τα σήμερα ισχύοντα χρηματοοικονομικά μέσα είναι ότι υπάρχει έτσι πολυσπερμία και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να, να, να, να επικεντρώσουμε τη στόχευσή τους για να είναι πιο διαχειρίσιμα. Κάτι άλλο τώρα το οποίο θα πρέπει να δούμε σε είναι με ποια κριτήρια και για ποιους στόχους θα πρέπει να θέτουν κάθε φορά πριν, προηγουμένως, για τα project τα οποία επιδέχονται ενίσχυση από αυτά τα μέσα. Αλλά έλεγχο και ενημέρωση και πληροφόρηση θέλουμε και πώς να είναι εδώ εμείς ως Κοινοβούλιο, ως Επιτροπή. Το για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρω Έχω κάποιε ερωτήσει, έχω κάποιε συμβολέ που να μου ξεκαθαρίσουν, γιατί έχουμε εδώ πέρα μια γνωμοδότηση 7 καθώς του Ελληνικού Συνεδρίου, όπου το συνέδριο επικρίνει την χρήση, τη λειτουργία τέλο πάντων αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων. Μπά και από αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μα διευκρινίσει. Θα βοηθούσε. Σε μια παραγραφή αυτή τη γνωμοδότησης τι λέει. Λέει ότι υπάρχουν κάποιε ανεπάρκειες για την κυκλική χρήση των πόρων, για το leverage ξέρω εγώ που θα μπορούσε να επιφέρουν αυτά τα μέσα και λέει ε, ε, τέλος πάντων ότι, ότι δεν δικαιολογείται η, ο τρόπος που αντιμετωπίζεται ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα και επίσης λέει εδώ πέρα ότι σε πολλούς τομείς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα. Και επίσης αναφέρεται η γνωμοδότηση και ο περιορισμός της στήριξης σε κάποια τέτοια συμβατικά μέσα πολιτικής οικονομικής και να μην χρησιμοποιούμε τα derivatives και, τα άλλα τα δομημένα ομόλογα τα οποία είναι οίκιστα διαφανή μέσα. Τι γίνεται εδώ, γιατί το λένε αυτό, γιατί τα φοβούνται, ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούν. Γιατί τα λέει αυτό το ελληνικό συνέδριο, άρα θα ήταν χρήσιμη η απάντηση της Κομισιόν. Εδώ θα βάζω τελεία, αλλά θα τα ξαναπούμε. Είναι σημαντικό το θέμα και ενδιαφέρον για την Επιτροπή μας, αλλά και για όλη την Ένωση. Γιατί μέσω αυτών των χρηματιστηριακών εργαλείων θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε αυτά που χρειαζόμαστε, τα έργα υποδομής και λοιπά, για να πάμε στην ανάπτυξη που θέλουμε. Όχι και όχι μόνο με τον κοινοτικό ή τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Αιδέρ, πράγματι. Πρέπει να προσπαθήσουμε με μια καλύτερη διευκρίνηση του τι σημαίνει χρηματοπιστωτικό μέσο δεν ξέρω τώρα αν αυτή η έννοια υπάρχει, έχει την ίδια απόχρωση σε όλες τις ε, γλώσσες, αλλά σε πολλές γλώσσες έχει μια αμφισημία. Μιλάμε για χρηματοπιστωτικές ε, προοπτικές, γαλλικά όταν λέμε φινανσίε εννοούμε ή δημοσιονομικό ή χρηματοπιστωτικό. Και όταν μιλάμε εδώ για καινοτόμα εργαλεία είναι καινοτόμα εργαλεία στον τομέα του προϋπολογισμού ή της, ε, του χρηματοπιστωτικού τομέα ή αναμειγνύουν και τα δύο, υπάρχει μια μία Και αυτή η έκθεση είναι και μια ευκαιρία να διευκρινίσουμε καλύτερα και την έννοια και το περιεχόμενο, τον τρόπο λειτουργίας, τους στόχους, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια. Έχουμε λοιπόν ζητήσει να γίνει μια μελέτη όπου θα υπάρξει και μια παρουσίαση τον επόμενο μήνα και όπως το υπενθύμησε η ΕΙΔΕΡ χρονοδιάγραμμα είναι παρουσίαση μιας έκθεσης γραπτής από την εισηγήτρια στις 31 Μαΐου. 12 Ιουνίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Η Οικονομική Επιτροπή και η Βιομηχανική Επιτροπή θα εγκρίνουν την έκθεσή τους μέσα στον Ιούνιο. Η τελική μας έκθεση θα έρθει τον Ιούνιο. Θέλεις να με διορθώσεις, ναι, πράγματι. Η προθεσμία για τις είναι 21 Ιουνίου και όχι 12 Ιουνίου. Ναι, είναι 12 γιατί είναι το αντίστροφο του 21. Η Αίντερ είναι συμβολίστρια και διάλεξε την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου. Πρέπει να τη σεβαστούμε. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 8 που είναι η έκθεση Γκάιερ για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εκεί είναι. Ναι, ναι, Άιντερ, έχεις το λόγο. Δεν θέλω να μονοπολίσω τη συζήτηση, αλλά είχα θέσει και ένα ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν μπορεί να απαντήσει. Μπορεί να απαντήσει η Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Εν συντομία μπορώ να σας πω ότι το ελεγκτικό συνέδριο στην έκθεσή του αναφέρεται στην επιμερισμένη διαχείριση, δηλαδή κυρίως στα θέματα της πολιτικής συνοχής. Ενώ η πρόταση της Κομισιόν για τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία και τις πλατφόρμες τους αφορά την άμεση ή έμεση διαχείριση από την Κομισιόν, είναι δηλαδή εκτός της σφαίρας της επιμερισμένης διαχείρισης. Ως εκ τούτου προτείνω να αποσταλεί στην κυρία και στη Γραμματεία ένα έγγραφο εργασίας της Κομισιόν, το οποίο νομίζω ότι δίνει απάντηση σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έθιξε το ελεκτικό συνέδριο και επί τη βάση αυτή μπορούμε να έχουμε μια άτυπη ανταλλαγή απόψεως στην Επιτροπή Προϋπολογισμών εφόσον το επιθυμεί. Πολύ ωραία, τρέμπια λέει ο πρόεδρος. Τούτο έχω των πραγμάτων, περνάμε στον κύριο Γκάιερ. Έχετε το λόγο. Και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ευχαριστώ. Έχω κρυφτεί εδώ πέρα. Τέρμα δεξιά, εδώ, εδώ είμαι. Βεβαίω καλό θα ήταν η Κομισιόν από το έγγραφο εργασίας να βάλει τα σημεία εκείνα τα οποία συμπεριέλαβε στην απόφαση περί απαλλαγής ε, την έκθεση Φιέλνερ δηλαδή το Κοινοβούλιο. Για να μην καθυστερούμε κιόλα. Λοιπόν, τώρα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σε μια προηγούμενη συνεδρίαση ήδη μιλήσανε ε, με βάση κάποιες ιδέες που είχα παρουσιάσει Μιλήσαμε λοιπόν για το ότι δεν είναι πολύ επίμαχο το θέμα αυτό. Γι' αυτό ελπίζω να συμφωνήσετε με τις προτάσεις ε, που έχω υποβάλει εδώ πέρα επί των προτάσεων της Κομισιόν. Απέσυρα τις τροπολογίες 16, 18, 19 και 20, την αξιολόγηση δηλαδή του προγράμματος για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θα ήθελα να έχω τουλάχιστον ένα, μια λύση έτοιμη. Να σας υπενθυμίσω πως θέλουμε να προωθήσουμε τέσσερις θεματικούς στόχους. Κινητικότητα εργαζομένων, ε, καταπολέμηση της φτώχειας, κοινωνική ενσημάτωση και θεσμική η ικανότητα και αποτελεσματικότητα της δημοσίας διοίκησης. Ξέρουμε πως αυτά είναι καλά, καλές επενδύσεις και βεβαίω θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε εκείνες τις διοικητικές ικανότητες που βρίσκονται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές ή όταν πρόκειται για κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων, 20% των κονδυλίων θα πάει σε κοινωνική ενσωμάτωση, τουλάχιστον 20% κοινωνική ενσωμάτωση κατά πολέμηση στόχιας και παρεμβάσεις ε, προτεραιότητας, όπως λέμε σε ωραία γερμανικά. Όσον αφορά τώρα τους τρεις τομείς που προτείνει η Κομισιόν, δηλαδή λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, θα πρέπει τουλάχιστον να πάνε εκεί πέρα 25% των διαρθρωτικών ταμείων μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Με τα νούμερα που ξέρουμε 40,7 δισεκατομμύρια και θα πρέπει να πάει ένα 40% στο Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 50 δισεκατομμύρια και βεβαίως για τις λιγότερα αναπτυγμένες περιοχές το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα είναι ε, το μεγαλύτερο κομμάτι των πληρωμών, 52% ε, δηλαδή 27, 27 ε, δισεκατομμύρια συνολικά. Μετά από την πρώτη συζήτηση κατέθεσα, περιορίστηκα σε κάποιες οριζόντιες ε, τροπολογίες που ελπίζω να αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας γιατί τα συζητήσαμε ούτως ή άλλως τα κείμενα με τους συντονιστές και περιορίζομαι σε ελάχιστες προτεραιότητες. Ενίσχυση του έκτος μέσου, το να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις και να έχουμε καλύτερο συντονισμό με άλλα προγράμματα για καινοτομία, απλοποίηση της χρηματοδότησης, επίσης να υπάρξουν κατά αποκοπήν χρηματοδοτήσεις για διοικητική απλούστευση. Γνωρίζουμε όλοι τα παράπονα που υπάρχουν για σοβαρή γραφειοκρατία, υπερβολικές ε, απαιτήσεις και διατάξεις, οπότε οι πληρωμές αυτές ε, κατά θα πρέπει να δημιουργήσουν μια πρώτη βελτίωση και βεβαίως να υπάρξει νέος ορισμός της ενεργείου ενσωμάτωσης ε, στους ε, ορισμούς. Αυτό το οποίο δηλαδή ζητάνε στην άλφη από την Επιτροπή Απασχόλησης αντί για τον πιο λιτό ορισμό της Κομισιόν. Αυτά και αναμένω τους αποθετήσεις σας. Très σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν σχόλια. Ο κύριος Κοσλόφσκι. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκάιερ για την γνωμοδότησή του, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι μια πρόταση την οποία τη χαιρετίζω. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι χρειάζεται να υπάρξει καλύτερο συντονισμό των πολιτικών και χρειαζόμαστε και σαφείς οριοθετικές γραμμές μεταξύ του χώρου, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Ανάπτυξης, του Αγροτικού Ταμείου για να μην υπάρξουν προβλήματα επικαλύψεων και να έχουμε το καλύτερο επίπεδο αποτελεσματικότητος. Πρέπει να είναι λοιπόν καλά κατευθυνόμενο το, το ταμείο αυτό και γι' αυτό ζητώ να υπάρξει και πρόταση από την Κομισιόν για την απλοποίηση της λειτουργίας του Κοινωνικού Ταμείου. Η ιδέα του πρότυπου μοναδιαίου κόστους και η καταποκοπή αντιμετώπιση νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι θετικό και συμφωνώ με τον κύριο Γκάιρο ότι τα κάτι μελη θα πρέπει αυτά να προχωρήσουν σε μια <clears throat> απλοποίηση και να σταματήσουν να την εμποδίσουν. Και επίσης χαίρομαι και για την πρόταση να υπάρξουν αποτελεσματικοί δείκτες για τα προγράμματα αυτά. Πιστεύω ότι η Κομισιόν θα μπορούσε να λάβει υπόψη και την ε, προσθέμενη αξία των συνολικών χορηγήσεων και τα αποτελέσματα τα οποία προσπορίζονται οι αποδέκτες. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για να χρησιμοποιήσουμε και το δυναμικό των νέων και των αναπήρων που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Είμαστε σε χαλεπούς καιρούς στην Ευρώπη και ιδίω για τι ευπαθεί αυτέ ομάδε που ανέφερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν πρόκειται να εξαλείψει την ένδια και την ανεργία μόνο του. Με μια καλή όμω διαχείριση μπορεί πράγματι να συμβάλλει <clears throat> στο να προωθηθούν στρατηγικές οι οποίες θα οδηγήσουν και στην ε, σωστή χρησιμοποίηση των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μα με τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων, με το να ε, μην υπάρξουν προσκόμματα και εμπόδια για μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Σας ευχαριστώ αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Η προθεσμία τροπολογιών είναι 16 Μαΐου στις, ε, το μεσημέρι. Θα υποβάλουμε λοιπόν στις 20 Ιουνίου, θα ψηφίσουμε την έκθεση του κύριου Γκαϊέρ. Η Επιτροπή απασχόλησης στις 10 Ιουλίου θα ψηφίσει και η ημερομηνία για την Ολομέλεια ακόμα δεν είναι απόλυτα γνωστή. Αυτά για το σημείο 8. Έχουμε ένα λουκούμιο σημείο που είναι το σημείο υπαριθμών 9, αλλά δεν είναι παρόλο εισηγητής. Θα τον αντικαταστήσω εγώ όμως. Σχέδιο <clears throat> κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης για την Λιγουρία και την Τοσκάνη μετά από τις πλημμύρες του προηγούμενου Οκτώβριου. Η Κομισιόν έχει παρουσιάσει μια πρόταση χρησιμοποίησης του Ταμείου αυτού και μια πρόταση μεταφοράς πιστώσεων ως ήθιστε για να χρηματοδοτηθεί αυτή η κινητοποίηση είναι ο διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 2 που έχει ήδη γίνει δεκτός από την Κομισιόν στι 6 ε, Μαρτίου. Οι ζημίε αυτών των πλημμυρών είναι τη τάξη και παραπάνω 700 εκατομμύρια ευρώ λόγω βλάβη σε υποδομέ σε δημόσιε μεταφορέ, σε στεγάσεις, σε επιχειρήσεις και πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Το Συμβούλιο θεωρεί λοιπόν ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το πρωτόκολλο 1 ε, για τη, στην συνθήκη της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να υπάρξουν 8 περαιτέρω εβδομάδες για να περιμένουμε τις, ε, τα σχόλια των Εθνικών ε, Κοινοβουλίων, ώστε η επιστολή αυτή προς την Κομισιόν θα εγκριθεί μάλλον στις 30 Μαΐου. Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν Θα μπορούμε λοιπόν στη συνέχεια να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν είναι καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες 29 Μαΐου. Η Επιτροπή Περιφερειακών Επιθέσεων θα μας δώσει τη γνωμοδότηση στις 30 Μαΐου και μετά στην επόμενη συνεδρίασή μας θα μπορούμε να ψηφίσουμε για την έγκριση στις 12 και 13 Ιουνίου. Εάν δεν υπάρχουν πόσες σχόλια, σας ευχαριστώ. Είμαστε στο τελευταίο σημείο της ημερία διάταξης, buildings policy, πολιτική ακινήτων. Θυμάστε ότι την ε, Δευτέρα η Μόνικα Χολμάιερ μας παρουσίασε το πρόβλημα εκείνο το οποίο αφορούσε το κτίριο Eastman σε σχέση με το σπίτι της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αποφασίσαμε να γνωμοδοτήσουμε σχετικά και αυτό θα γίνει στις 31 Μαΐου. Επομένως, κλείσαμε και αυτό, δεν έχουν τίποτα διάφορα, πέρασαν τριάδες.